Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινάμε τη συζήτησή μας, ε, ξαναξεκινάει η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της ε, χτεσινής συνεδρίασης ε, διανεμήθηκαν, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις, αν όχι εγκρίνονται τα πρακτικά. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, προβλέπει την παρουσίαση του Συμβουλίου τη θέση του για το Γενικό Προεπολογισμό του 2013. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο ευθύς αμέσω στον κύριο Μαυρογιάννη Ανδρέα που θα μιλήσει εξ ονόματος Συμβουλίου. Παρακαλώ κύριε Μαυρογιάννη. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού που αφορά το οικονομικό έτος 2013. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν ήξερα ότι πρέπει να είμαι όρθιος. Το ξέχασα. Ξέρετε μετά από τι καλοκαιρινές διακοπέ, κάποια πράγματα τα ξεχνάει κανεί Καλό είναι να μα τα υπενθυμίζουν και να μα επαναφέρουν στην πραγματικότητα. <clears throat> για μια ακόμα φορά θέλω να τονίσω ότι είναι για μένα μια μεγάλη τιμή που μπορώ να σα παρουσιάσω τη θέση του Συμβουλίου σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2013 όπω έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο στι 24 του Ιουλίου του 2012 είναι φυσικά διατεθειμένο το Συμβούλιο να συνεργαστεί τόσο με το Κοινοβούλιο όσο και με την Κομισιόν κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και μηνών ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία <clears throat> σε σχέση με ένα εξισορροπημένο και ρεαλιστικό προϋπολογισμό για το 2013. Έχω κάθε πεποίθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό εάν υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ μας. Το Συμβούλιο από τη δική του πλευρά είναι απόλυτα έτοιμο να εργαστεί επικοδομητικά και με πνεύμα συμβιβασμού για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Ο πρώτος τριγωνικός διάλογος για τον προϋπολογισμό έλαβε χώρα στις 9 Ιουλίου, είχε θετικό χαρακτήρα και ήταν ενθαρρυντικός. Στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις προτάσει της Κομισιόν και το Συμβούλιο στάθμισε τη θέση του για το 2013 και προβλέπει μια αύξηση κατά 1,27% σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 2,79% σε πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στους, στα τρία σημαντικά σημεία τα οποία διατρέχουν τη θέση του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο αποφάσισε να αποδώσει προτεραιότητα σε προγράμματα και δράσεις του προϋπολογισμού που θα βοηθήσουν την έξοδο από την τωρινή οικονομική κρίση, θα υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση των οικονομιών, θα δημιουργήσουν μόνιμες ευκαιρίες και θα παροτρύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, επειδή το 2013 είναι το τελευταίο έτος του τωρινού δημοσιονομικού πλαισίου, <clears throat> το Συμβούλιο πρότεινε μια αύξηση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που ξεπερνάει σημαντικά το επίπεδο του πληθωρισμού. Τρίτον, το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη τα μέτρα τα οποία έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη για την εξυγίανση των εθνικών τους προϋπολογισμών και μέσα στο τωρινό οικονομικό κλίμα έχει αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο να παραμείνουν υπό οι διοικητικές δαπάνες ακολουθώντας και την ε, εγχώρια πολιτική των κρατών μελών. Θα διεξέλθω τώρα τα κύρια στοιχεία της θέσης του Συμβουλίου για κάθε μία από τις επικεφαλίδες και υποεπικεφαλίδες του Δημοσιονομικού Πολιετούς Προγράμματος. Ξεκινώ με την επικεφαλίδα 1, βιώσιμη ανάπτυξη. Το Συμβούλιο εδώ θεωρεί ότι αυτή η επικεφαλίδα θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις πρώτες προτεραιότητες στον προϋπολογισμό του 2013. Για το λόγο αυτό έχει προτείνει μία σημαντική αύξηση τόσο σε πιστώσεις υποχρεώσεων ως κατά 2,79% όσο και σε πιστώσεις πληρωμών κατά 6,71%. Η αύξηση αυτή θα εξασφαλίσει ότι υπάρχει η επαρκής χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να, εφαρμοστεί το σύμφωνο για την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση που αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και δράσεων που εμπίπτουν σε αυτή την επικεφαλίδα και που διαδραματίζουν κέριο ρόλο στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θα οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και επίσης το Συμβούλιο έχει εργαστεί για να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τις διαρτωτικέ δράσεις. Στην υποεπικεφαλίδα 1β, συνοχή για την ανάπτυξη και την ε, απασχόληση, οι πιστώσεις πληρωμών θα αυξηθούν κατά πάνω από 8% έναντι του 2012. Σε σχέση με την επικεφαλίδα 2, διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων, το Συμβούλιο προτείνει μια σταθεροποίηση του επίπεδου πιστώσεων υποχρεώσεων σε σχέση με το 2012. Αλλά λόγω της επιταχυμένης εφαρμογής στο τελικό έτος των πολιετών, των τρέχουσών πολιετών προοπτικών υποστηρίζει μια αύξηση κατά 440 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών έναντι του 2012. Οι περικοπές που εφαρμόζονται σε αυτή την επικεφαλίδα είναι αποτέλεσμα μιας ανάλυσης της ε, εκτέλεσης των προηγουμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού και της προσδοκόμενης ικανότητας απορρόφησης. Βασίζονται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη θέση μας και υπόκεινται σε αναθεώρηση μετά από την παρουσίαση από τη βλάβη της Κομισιόν της παραδοσιακής επιστολής για διορθωτικό προϋπολογισμό στο φως του αγροτικού έτους 2012. Επικεφαλίδα 3. Πολίτες, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Εκεί το Συμβούλιο υποστηρίζει με τριοπαθείς περικοπές και σε πιστώσεις πληρωμών και σε πιστώσεις υποχρεώσεων, διότι θεωρεί ότι η αύξηση η οποία προτινόταν από την Κομισιόν θα ξεπερνούσε τη ρεαλιστική ικανότητα απορρόφησης για τα μέτρα αυτά. Μόλον τούτο το Συμβούλιο έχει προτείνει μια σημαντική αύξηση 5% σε πιστώσεις πληρωμών για την υποεπικεφαλίδα 3α που είναι η ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη με στόχο να ενισχύσει διάφορες γραμμές του προπολογισμού και ιδίω τη γραμμή του προπολογισμού που έχει να κάνει με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Σε ό,τι αφορά την επικεφαλίδα 4, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτη το Συμβούλιο έχει θέσει τις πιστώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων στο χαμηλότερο επίπεδο που ζήτησε η Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη και τρέχουσα εκτέλεση και απορρόφηση του προπολογισμού και τις ρεαλιστικές προσδοκίες απορρόφησης και επίσης και τις απαιτήσει που χρειάζονται σε διάφορα χρόνια του προπολογισμού. Αυτή η κατηγορία μαζί με την υποκατηγορία 1α και 1β και 2 καλύπτεται από μια δήλωση για πιστώσεις πληρωμών όπου το Συμβούλιο προσκαλεί την Κομισιόν να υποβάλει ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αν οι πιστώσεις πληρωμών του 2013 ξεπεράσουν τις προβλεπόμενες ανάγκες. Για τον τομέα 5, διοικητικές δαπάνες. Το Συμβούλιο, ως ήθιστε, δεν έχει τροποποιήσει το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού, ενώ το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την Κομισιόν και άλλα θεσμικά όργανα για να μειωθεί η αύξηση στο διοικητικό του προϋπολογισμό, έχει εντοπίσει περαιτέρω δυνατότητες εξοικονόμησης και ως εκ τούτου έχει θέσει τις διοικητικές, τα διοικητικά κονδύλια για την Κομισιόν και τα άλλα θεσμικά όργανα σε ένα επίπεδο πολύ κοντά από το επίπεδο του 2012. Το Συμβούλιο επίσης έχει απορρίψει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα οργανογράμματα των θεσμικών οργάνων εκτός από τις θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την προσχώρηση της Κροατίας στο φως της πρότασης της Κομισιόν να υπάρξει μείωση κατά 5% του αριθμού των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα 2013-2017, το Συμβούλιο έχει εφαρμόσει μια μείωση κατά 1% στο οργανόγραμμα των θεσμικών οργάνων πέραν της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης λόγω της πρόσφατης δημιουργίας της και επίσης και στην, με την εξαίρεση του Ευρωπαϊκού Επόπτη δεδομένων και του διαμεσολαβητή λόγω του μικρού μεγέθους των δύο αυτών φορέων. Τέλο, ό,τι αφορά του αποκεντρωμένου φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει το επίπεδο κονδυλίων για του λειτουργικού προπολογισμού αυτών των φορέων, όπω προτείνεται από την Κομισιόν, κάτι το οποίο θα σημάνει αύξηση κονδυλίων κατά 1,98% κατά μέσο όρο, σχεδόν λοιπόν 2% μεσοσταθμικά από την ε, ε, ονομαστική, το ονομαστικό πάγωμα στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Επίσης, στις ήδη εδρεωμένες αποκεντρωμένες υπηρεσίες εφαρμόζεται η μείωση προσωπικού κατά 1%. Νέες θέσεις έγιναν δεκτές μόνο για φορείς που είναι στη φάση εκκίνησης ή των φορέων που έχουν αναλάβει νέα καθήκοντα. Γενικά το Συμβούλιο έχει αποφάσει <clears throat> να δεχτεί τη δημιουργία 185 νέων θέσεων στους αποκεντρωμένους φορείς πάνω από ένα τρίτο αυτών των θέσεων θα είναι για τις νέες χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές που εποπτεύουν τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις αγορές <clears throat> αξιογράφου. Κύριε Πρόεδρε και έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με το προϋπολογισμό του 2013 εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αναγνώρισης της δυσκολίας που υπάρχει στο οικονομικό κλίμα των κρατών μελών και της παροχής επαρκών κονδυλίων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υποστηριχθούν προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Στο σύμφωνο απασχόλησης και ανάπτυξης που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανέφεραν ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει καταλητικό ρόλο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Είναι η ελπίδα μου ότι αυτή θα είναι και η οδηγή γραμμή για όλου μα τι συζητήσει μα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2013 στι επόμενε εβδομάδε και μήνε, όσο προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του προϋπολογισμού του 2013. Σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, όλοι ο πρόεδρος. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Λεβεντόφσκι. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητά μέλη, ε, η Επιτροπή, εγώ εξ ονόματος της ε, Επιτροπής έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τις ε, επιφυλάξεις μας όσον αφορά τον προπλογισμό του 2013 την ανάγνωσή του στο Συμβούλιο. Αυτά στα πλαίσια μιας ε, τριμερούς ε, στις 9 Ιουλίου και υπάρχει σχετική επιστολή του κ. Μπαρόζο προς τα κράτη-μέλη. Η ανάγνωση στο Συμβούλιο δεν είναι αντιφατική με ε, τα συμπεράσματα της, της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Έχουμε τα συμπεράσματα ε, των επιπτώσεων στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης και παραθέτω. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών συμφώνησαν ότι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει καταλήτη για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος της παράτασης Νομίζω ότι αυτό που προτάθηκε για το 2013 είναι συμβατό με τη λογική που διέπει ε, αυτή την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Πιέζουμε προς τα κάτω τις ε, δεσμεύσεις, αλλά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ε, σε πάρα πολλούς τομείς να μπορούμε να αυξήσουμε τους ε, τομείς ε, για την ε, ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Το πρόβλημα είναι οι δαπάνες. Στο τέλος των δημοσιονομικών προεπτικών δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Αλλά αυτό δεν εκπλήσει κανένα. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις επενδύσεις σε πάρα πολλά κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός του 2011 ήταν ήδη πολύ συρρυκνωμένος, τουλάχιστον κατά 5 εκατομμυρία, χαμηλότερος κατά 5 δισεκατομμύρια και αυτό ε, δεν μας ε, βοήθησε στο να επιτύχουμε την ε, δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη-μέλη. Έχουν αυξηθεί οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις. Εμείς προτείναμε μια αύξηση της τάξης του 6,8% αλλά αυτό στον τομέα της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των θέσεων απασχόλησης. Εκείνο που έχει σημασία, ανεξάρτητα αν, αν έχουμε δίκιο ή λάθος, είναι ότι όσον αφορά την ανάπτυξη για εφέτος, μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 9 δις κατά 9 δις μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι πέρυσι. Και πέρυσι είχαμε ήδη έλλειψη κονδυλίων για επιστροφή. Τώρα λοιπόν έχουμε εξαντλήσει πλήρως τα κοινωνικά ταμεία και το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης ε, που αφορά ε, τις περισσότερο αναπτυγμένες ε, περιοχές της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι σωστό είναι αυτό να αυξάνονται τα αιτήματα για καταβολές κυρίως σε περιοχές που συμβάλλουν ε, στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να πω για άλλη μια φορά ότι απογοητεύτηκα από το το Συμβούλιο περιέκοψε τις υποχρεώσεις κατά 5 δις ευρώ και οι μεγαλύτερες περικοπές έγιναν στον τομέα 1α. Ε, πρόκειται για τον τομέα που αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό όμως αφορά και τη συνοχή. Και όσον αφορά στη συνοχή, ε, στο Συμβούλιο υπάρχει μια παραδοχή σχετικά με την πολύ κατηστορημένη εκταμίευση στα κράτη-μέλη. Αυτά όσον αφορά την αλληλεγγύη μας ε, προς τους εταίρους μας ανά τον κόσμο. Τίθεται επίσης και το θέμα των διοικητικών περιορισμών. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο βαθμό του δυνατού. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι εις βάρος της αποτελεσματικότητας της διοίκησης που έχει αναλάβει πλέον πολύ μεγαλύτερα καθήκοντα από ό,τι κατά τα προηγούμενα έτη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς μπορούμε ρεαλιστικά να καθορίσουμε ε, ικανοποιητικά επίπεδα πληρωμών ε, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Και είμαι ευγνώμων στα μέλη του Συμβουλίου και στον κύριο Λαμασούρ για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν να συζητήσουν ποια είναι τα κριτήρια και τα σημεία αναφορά, έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιοπρεπέ επίπεδο καταβολών ε, πληρωμών, όχι υπερβολικό, αλλά να μπορούμε εν πάση περιπτώσει να ε, καταβάλουμε τα χρήματα που είναι απαραίτητο. Και πριν από την ολοκλήρωση τη συνδιαλλαγή, πρέπει να υπάρχει βούληση να γνωρίζουμε γνωρίζουμε ποιε είναι οι δημοσιονομικέ προοπτικέ, ε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μα τι αποφάσει που έλαβαν τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο, στον κύριο Σαλβαδόρ Πογέδο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Συμβούλιο για την παρουσία του και τις εξηγήσεις που έδωσε για τον προϋπολογισμό του 2013. Φαίνεται στοιχειώδες, πολλές φορές όμως στο παρελθόν δεν είχε προσέλθει το Συμβούλιο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο ε, που παρουσιάζει τη θέση του παρά το γεγονός ότι πολλές φορές φαίνεται ακατανόητη η θέση του Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο. Οι στόχοι μας είναι κοινοί, να αντιμετωπίσουμε την κρίση, να ευνοήσουμε την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν έχει κάνει την εργασία της, την έχει κάνει σωστά, με έναν τρόπο συνεκτικό και συνεπή. Δεν έχει νόημα να διευρύνουμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων όταν δεν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις πληρωμών. Η Κομισιόν θέλει να μειώσει τα λεγόμενα ραλ, τα υπόλοιπα τα οποία έχουν απομείνει, τα οποία ήδη έχουν μεταφερθεί από το προηγούμενο προϋπολογισμό στο 2012. Γνωρίζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου τα προβλήματα που έχουν τα υπολείμματα αυτά τα οποία φτάνουν ουσιαστικά σε επίπεδο ενός ετήσιου προπολογισμού. Δεν καταδεικνύουν αυτά τα υπολείμματα υποχρεώσεων την, ε, δεν υπονομεύουν την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλουν οι πολίτες που θέλουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική συγχρόνως. Υπάρχει πάντα η παραδοσιακή αυτή στάση του Συμβουλίου να κάνει γραμμικές ε, μειώσεις για να προσαρμόσει τις προβλέψεις του προπολογισμού στις πιέσεις που ασκούνται από τα κρατημέλη. Μια τέτοια αντιμετώπιση όμως θα πρέπει να ανήκει στην ιστορία. Δεν βοηθάει κανένα γιατί πάνω απ' όλα οδηγεί σε μια στρέβλωση της σωστής χρήσης των πόρων του προπολογισμού που είναι διαθέσιμες. Το να βγάλουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνονται επί τη βάση των προβλέψεων που αστέλνουν τα ίδια αυτά κράτη-μέλη σε σχέση με την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού αυτό θα έχει παράπλευρα αποτελέσματα που είναι φανερό ότι θα είναι αρνητικά. Πρέπει κύριε Πρόεδρε να συγκεράσουμε την λιτότητα με το ρεαλισμό. Πάντα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν δει τον προπολογισμό του Συμβουλίου με έναν τρόπο θετικό. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ τη λιτότητα που θίγει τα κράτη-μέλη και της ανάγκης ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί περιμένουμε μεγαλύτερη <clears throat> ευκαμψία και πιο ευρωπαϊκό πνεύμα. Το περιμένουμε από όλου του εμπλεκομένου. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ακόμα και αν είναι διαφορετικέ ασκήσει προπολογισμού, ο προπολογισμό του 2013 και οι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ συνδέονται άρρηκτα και λόγω τη χρονική του συνάφεια και λόγω του γεγονότο ότι δεν θα απαιτήσουμε στο μέλλον άλλε ε, αναλήψει υποχρεώσεων όσο χρειαζόμαστε χρήματα για να κλείσουμε τα τωρινά υπόλοιπα. Ευχαριστώ κύριε Γκαρίγα. Δίνω το λόγο στον κύριο Τζοβάνι Λαβία, ο οποίος είναι εισηγητής για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ε, κύριε Λεβαντόφσκι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου για τον προεπλογισμό του 2013 κατιστά σαφές ότι υπάρχει μια ουσιαστική αντίφαση ανάμεσα σε αυτό που είπαν στις 28 και στις 29 Ιουνίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και σε αυτό που αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Από τη μια μιλάνε για επενδύσεις για την ανάπτυξη, ε, την απασχόληση και από την άλλη όμως ενώ προβλέπεται να γίνουν μεγάλες ε, περικοπές ε, κυρίως εκείνες τις γραμμές του προεπλογισμού που χρηματοδοτούν τις ε, σχετικές πολιτικές ακριβώς για να δημιουργηθεί η ανάπτυξη και οι θέσει απασχόλησης κυρίως για τους νέους Ευρωπαίους όπως ε, είχα την ευκαιρία να πω και σε άλλες, περιπτώσει, ε, περιπτώσεις γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες τις οικονομικές που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη στο εσωτερικό τους όμως η απάντηση στην κρίση όπως εξάλλου φάνηκε από το Συμβούλιο σε δημόσιες δηλώσεις του δηλαδή σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο η απάντηση είναι περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Άρα δηλαδή δεν είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα εκ των προτέρων να ορίζουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πληρωμών, όπως θα έκανε το Συμβούλιο, που είναι σαφώς χαμηλότερο. Μιλάμε για μια περικοπή πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπαν οι προαλήσαντες, από τα στοιχεία, από το ποσό εκείνο που θεώρησε η Κομισιόν ότι είναι απαραίτητο για να διαφυλαχθεί ο προπολογισμό. Θα ήθελα να στον πρόεδρο του Συμβουλίου ότι το ποσό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προέκυψε από τις εκτιμήσεις που έκαναν τα κράτη-μέλη. Και αυτά όμως αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω από τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν, ε, όσον αφορά τις ανάγκες ε, του προϋπολογισμού, όπου αναφέρεται η αύξηση του 6,8 σε σχέση με τον προπολογισμό του 2012, αυτό το ποσό δεν είναι αυθαίρετο. Είναι μια ρεαλιστική αξιολόγηση των κονδυλίων που είναι απαραίτητα και που την έκανε η Επιτροπή με βάση τα στοιχεία που κατέθεσαν τα κράτη-μέλη. Και αυτό το για να ικανοποιήσουμε και να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Εξάλλου δεν είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα να διατρέξουμε κίνδυνο, να προκύψει κίνδυνο στο να μπλοκαριστούν συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν χρήματα ο ίδιος ο πρόεδρος κύριος Μπαρόζο έκρινε ότι είναι σκόπιμο να αποστείλει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων μια επιστολή όπου θα εκφράζει τις ανησυχίες του για τις οριζόντιες περικοπές. Νομίζω δεν είναι υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει με τη βοήθεια της Επιτροπής να αποκτήσει τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στις πληρωμές του 2012. Ελπίζω ότι η διοργανική ε, συνάντηση στις 26 Σεπτεμβρίου θα αποδειχθεί ότι θα είναι χρήσιμη για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες και για να αποδείξουμε όλα αυτά τα δυσάρεστα που έχουν λάβει η χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι για να πλησιάσουμε τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και για να υπάρχει μια υπεύθυνη ανάγνωση που θα διασφαλίζει ότι ε, ο προϋπολογισμός είναι προστασμένος σε ανάπτυξη, ε, πρέπει να λάβουν όλα αυτά υπόψη αυτά που ελέγχθησαν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαβία και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Μπόγκαν ε, που είναι ο εισηγητής του Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, ως εισηγητής θέλω να εστιάσω την προσοχή μου στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους άλλους τομείς του προϋπολογισμού Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε λάβει υπόψη την επιστολή που απεστάλλει από τον Επίτροπο κ. Λεβαντόφσκι στην αρχή του χρόνου ζητώντα από τα θεσμικά όργανα να διατηρήσουν τις αυξήσεις του διοικητικού του προϋπολογισμού κάτω από το 1,9%. Νωρίτερα εφέτος το Κοινοβούλιο μας αποφάσισε μια αύξηση κατά 1,9% το 2013 πέραν του πρόσθετου κόστους που εκνομιζόμαστε λόγω Κροατίας. Παγώσαμε και πάλι όλα τα επιδόματα των βουλευτών και αποφασίσαμε να μειώσουμε τον προϋπολογισμό ταξιδιών κατά 5% και θεσπίσαμε και μια σειρά από άλλα μέτρα για εξοικονομήσεις. Νωρίτερα λοιπόν το έτος όταν συζητούσαμε την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίσαμε ότι περιμέναμε να υπάρχουν περισσότερες εξοικονομήσεις το φθινόπωρο. Ο στόχος θα ήταν να έχουμε 1,9% αύξηση αλλά συμπεριλαμβανομένη και της Κροατία. Οι περισσότερε άλλε πολιτικέ ομάδε συμφωνούν με κάτι τέτοιο και του ευχαριστώ για τη συνεργασία του. Για να πετύχουμε όμω αυτό το στόχο του 1,9% μαζί με την Κροατία πρέπει να βρούμε άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήσεων από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοίταμε τώρα ποιε είναι οι δυνατότητε για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Εάν πράξουμε όμω κάτι τέτοιο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη να κάνουμε εξοικονομήσεις αλλά συγχρόνως να μην γίνονται εξοικονομήσεις που θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου μας και την αποτελεσματικότητα των μεμονωμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πω και κάτι για τους άλλους τομείς του προπολογισμού και άλλα θεσμικά όργανα δέχτηκαν να παραμείνουν στα πλαίσια του 1,9% παρά την προσχώρηση της Κροατίας και του 1,5 για τις αυξήσεις των αποδοχών των υπαλλήλων. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προέβλεπε μια αύξηση κατά 10% και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είχε ζητήσει μια αύξηση μεγαλύτερη από 1,9% γιατί είπε ότι είναι νέο θεσμικό όργανο με νέες ευθύνες ιδίως στον τομέα της ασφάλειας. Γι' αυτό αντί να έχουμε μια ένα συλλήβδεν πάγωμα των κονδυλίων θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε θεσμικού οργάνου πρωτού αποφασίσουμε ποια θα πρέπει να είναι η αύξηση και περιμένω ότι και το Συμβούλιο θα αποδηθεί σε αυτό το εγχείρημα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν και τα περισσότερα θεσμικά όργανα θα έχουν μια αύξηση τη τάξη του 1,9% όπως πρότεινε η Κομισιόν. Αυτά είναι καλές ειδήσει καταδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη αναγνωρίζουν τις χρηματοοικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζουμε και είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε με τρόπο ο οποίος είναι υπεύθυνο. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι και μετά στο Συμβουλίο στον κύριο Μαπρογιάννη. Παρακαλώ κύριε Λεβαντόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ χαιρετίζω τις παρατηρήσεις του Σαλβαδόρ από και αυτά τα οποία ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Λαβία καθώ και ο κύριο Βόγκαν Έχουμε ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για να καταλήξουμε σε μια σωστή χρηματοδότηση για την Ευρώπη το 2013 ακολουθώντας και τις αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ζήτησαν να υπάρξουν επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το Συμβουλίο υπό την ηγεσία του Ανδρέα Μαυρογιάννη έχει δείξει ότι είναι έτοιμο να εμπλακεί σε ένα διάλογο για έγκαιρη συμφωνία. Επομένως, για να έχουμε πραγματικές προοπτικές αναπτύξεως και επενδύσεων το 2013. Ευχαριστώ κύριος Μαυρογιάννης για το Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάγη Γαπολέδο, τον κύριο Λαβία, τον κύριο Βόγκαν για τα πολύ επικοδομητικά σχόλιά τους και θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Επίτροπο κ. Λεβεντόφσκι για τα σχόλιά του στο θέμα αυτό. Δεν βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ιδιαίτερα καρποφόρα αυτή η ανταλλαγή απόψεων, διότι καταδεικνύει ότι η παρουσίαση της θέσεως του Συμβουλίου για τον Σχέδιο Προϋπολογισμού του 2013 μας έχει επιτρέψει σε όλους μας να καταλήξουμε σε μια καλύτερη κατανόηση των θέσεων των μεν και των δε και υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για μια αμοιβαία συνέντευξη μεταξύ μας. Αυτή είναι η πρώτη απαράγραπτη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013 στους επόμενους μήνες. Και αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα στις προθεσμίες που θεσπίζουν οι συνθήκες. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι πρωταρχική σημασία να τηρήσουμε αυτέ τι προθεσμίε λόγω και των συνθήκων στι οποίε βρισκόμαστε. Η σημερινή συζήτηση ήταν ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για τη συζήτησή μα. Η διαδικασία του προπολογισμού Εφέτο λαμβάνει χώρα, όπω είπα προηγουμένω. σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Γι' αυτό πρέπει όλοι να εργαστούμε με επικοδομητικό τρόπο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε στο εγχείρημα αυτό και πρέπει να είμαστε και σε θέση να έχουμε ένα ρεαλιστικό και εξισορροπημένο προπολογισμό για το 2013. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου και εγώ προσωπικά, επειδή αναφέρθηκε σε μένα ο κ. Λεβαντόφσκι, αλλά εγώ είμαι απλώ ένα ταπεινό υπηρέτη σα στο θέμα αυτό, θα πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και συγχρόνω εγώ καταγράφω προσεκτικά το γεγονός ότι παραμένουν διαφορές απόψεων μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου και μεταξύ της θέσης του Συμβουλίου και των θέσεων που έχουν εκφραστεί από τα διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες σεβόμαστε. Ξέρετε ότι σεβόμαστε όλες τις εκφραζόμενες θέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Λεβαντόφσκι, είναι πρόθεσή μας μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν να προχωρήσουμε σε ένα τριγωνικό διάλογο στις 26 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουμε για το επίπεδο πληρωμών ήδη για το τρέχον έτος. Σε σχέση τώρα με τα σχόλια του κυρίου Λαβία, πιστεύω ότι στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά από τη δική μου εμπειρία, έχοντας συζητήσει διμερώς με όλα τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, όλοι, όλοι και οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να εξυπηρετεί στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να έχουμε μια ποιοτική εκτέλεση του προπολογισμού και να έχουμε καλύτερη δαπάνη των κονδυλίων. Βλέπω όμως να είναι κάπως μια ηρωνία αυτοί οι οποίοι θέλουν καλύτερη δαπάνη του προπολισμού να ζητούν συγχρόνως και περικοπές. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι δεν έχουν όλη την ίδια ερμηνεία του τι σημαίνει σωστή εκτέλεση του προπολογισμού. Υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση με την θέση του Συμβουλίου για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και ανάπτυξης και θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την αντίφαση και να εξασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο έχει διατηρήσει το συνολικό ποσό το οποίο θεωρήθηκε ότι ήταν διαθέσιμο το 2013, τα 55 δηλαδή δισεκατομμύρια από τα 120 εκατομμύρια του συνολικού προϋπολογισμού, γιατί είναι αυτό το ποσό το οποίο έχει σαν στόχο να εξυπηρετεί την ανάπτυξη. Θέλω να προσθέσω ακόμα ότι βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Κομισιόν τον παραδοσιακό της ρόλο ως έντιμο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και βασίζομαι ειλικρινά στις προσπάθειες του κυρίου Λεβαντόφσκι όπως και τα προηγούμενα χρόνια για να μας βοηθήσει να εξεύρουμε το σωστό δρόμο. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο Κοινοβούλιο στην εξέταση της θέσης του Συμβουλίου και προσβλέπω και στις διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο αλλά και Νοέμβριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαυρογιάννη. Έκλεισε η συζήτηση. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην κοινή συζήτηση ε, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερική πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Με, ε,